Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ. Επαλήθευση για την τροπολογία 10, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, Η κυρία Όμεν Ρόιτεν ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Yes, Πρόεδρε, καταλήξαμε σε συμφωνία με τους σκιώδεις εισηγητές για την προφορική τροπολογία για την παράγραφο 18. Αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία 26 και η παράγραφος 18 θα αποσυρθούν από την κυρία Φλότρ και άρα προτείνω στην ομάδα μου να υπερψηφίσει την τροπολογία 29 για αυτή την παράγραφο 18. Ευχαριστώ. Ε, okay. Ε, τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. 12? Για τη 12 τι σα είπα ότι απερίφθη. Ε, σωστά. Θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για το 12. Παρακαλώ. 12. 12. 12. 12. Επαλήθευση για το 12. Πέρας ψηφοφορίας. As I said, απορρίπτεται. Απορρίπτεται όπως έλεγα και προηγουμένως. Τροπολογία 29 υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, έχουμε μια... Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 26 και πάμε τώρα σε μια προφορική τροπολογία ε, επί της παραγράφου 18. Η κυρία Μενρόιτεν έχει το λόγο. Um, Μια προφορική τροπολογία θέλω να καταθέσω, να προσθέσω στην ε, παράγραφο 18 τα εξή, θα σας το διαβάσω. Ανησυχεί για την έλλειψη προόδου σε αυτές τις έρευνε και σημειώνει ότι η έσκατη κράτηση ε, γνωστών δημοσιογράφων όπως ο Νεντέμ Σενέρ και ο Άχμετ Σίκ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αξιοπιστία αυτών των φυλών που θα έπρεπε αντίθετα να ενισχύουν τη δημοκρατία. τροπολογία. Όχι. Άρα προχωράμε στην ψήφιση της παραγράφου 18 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Check 13. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Έλεγχος για την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Τροπολογία 3, check. Let's check on 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Like I said, εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Come on. 30. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 40 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 34 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 35 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Σήμερα είμαι διάθετος, οπότε το δέχομαι. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 5, παρακαλώ. Μόνο σήμερα είμαι διάθετος, πέρας ψηφοφορίας. What a surprise. Οποία έκπληξη, απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Check 18. Τη 18 επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας σοφορίας. Απορρίπτεται. 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Come again? Yeah, okay, yeah. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. You want to check what? 19? Τι 19 θέλετε ε, να ελέγξουμε. Είπα εγκρίνεται. 19 παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. 19. Πέρα σοφορίας. Ου. <laughs> Okay, I think the machines have a problem. Ε, έχει πρόβλημα το μηχάνημα. Δεν είναι σωστό το αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιος τεχνικός να έρθει να ελέγξει. Απερίφθη. 25 τώρα. Το 25. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Check. Check 25. 25 έλεγχος. Πέρας φοφορίας. Uh, ε, εγκρίνεται. Ε, ναι. We go to four. Τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Check number 4. Η 4. Επαλήθευση. Πέρας Βορείας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Check number 6. Πέρας οφορίας. Εγκρίνεται. 22 falls. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Okay, I need a win. I need a win, so we'll check nine. Πρέπει κάποιος να νικήσει. Έλεγχος για την εννέα, παρακαλώ. Πέρα οφορίας. Αχα. Απορρίπτεται. Final vote. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Ε, η επόμενη έκθεση. Διαδικασία ένταξης Μαυρομουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Check 1. Έλεγχος για την τροπολογία 1 παρακαλώ. Πέρας οφορία. Εγκρίνεται. Έκανα μία φορά ένα λάθος. Δεν σημαίνει ότι θα ασφάλω συνέχεια. Παράγραφος 32 σε δύο τμήματα. Πέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Γιαρόκα σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3 με ονομαστική κλήση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36 με ονομαστική κλήση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοβορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 41 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοβορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοβορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 98 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Was war's, Herr Präsident? Εγκρίνεται. Παράγραφος 100. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 102 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Γιώροκα. Τελευταία ψήφος για σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι. Έκθεση Λάγκε σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά Αποχές. Check 2. Επαλήθευση για τη 2 παρακαλώ. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. 3 ε, και 10 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 παράγραφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 51 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 54 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 59. Υπέρ. No. I'm sorry. Ναι, τροπολογία 5 στην παράγραφο 59. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 64 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Check. Paragraph 75. Παράγραφος 75. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Did I do paragraph 75? Yes, you did. No, no, no. that was for this one. Because you always have to, be very often have a Okay, my, my, my mistake, my mistake. Let's go back. Εγώ έκανα λάθος. Ε, γυρνούμε προς τα πίσω τώρα. Επιστρέφουμε στην τροπολογία 6. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 89 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 90 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος τροπολογία 9. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 108. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. 7. Την 7 έλεγχος παρακαλώ. Ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη F σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέλικη ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Σάλτη. Ακολουθούν τώρα οι επεξηγήσεις ψήφου.